Κύριε Εσταράς, θέλετε το λόγο από ό,τι κατάλαβα. Είναι διαδικαστικό. Έχουμε αεροπλάνα να πάρουμε. 11.30 ψηφίζουμε και καθυστερεί η ψηφοφορία. Καθυστερεί η συζήτηση γιατί απουσιάζει και η Επίτροπος και η Συγκήτρια. Ε, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά παρακαλώ να μην καθυστερήσουμε και να μην αναβάλουμε τις ψηφοφορίες για αυτό το λόγο. Έχουμε και ταξίδια. Το γνωρίζω το γεγονός ότι μας βλέπετε να καθόμαστε εδώ δεν σημαίνει ότι αδρανούμε. Επιλαμβανόμαστε. Εγώ δεν έχω άλλο τρόπο παρά να κάνω τηλεφωνήματα και επαφές, αυτό κάνουμε. Έρχεται η Επίτροπος. Ήρθε, είναι παρούσα. Έρχεται και η συγγήτρια. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Καθίστε παρακαλώ. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στην ε, εισηγήτρια. Ακόμα και από μπορούμε να ξεκινήσουμε. Commissioner, good morning. Uh, I would appreciate Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να αρχίσουμε. Έρχεται η συγκήτρια, αλλά